Ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα. Τα πρακτικά της ε, συνεδρίασης θα είναι διαθέσιμα σύντομα. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, τότε...